Hello everyone. Now we move to the session. Ωραία. Χαίρετε. Πρώτα απ' όλα να σας κάνω μια ανακοίνωση. Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες θέλω να ενημερώσω το Σώμα για τις εξή προτάσεις για αλλαγή στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης. Η συζήτηση για την προφερική ερώτηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων συμφωνίας ελευθερίου εμπορίου με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα καταλήξει με ένα ψήφισμα που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Την πρώτη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ο κύριος Σόλτς.